Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε Νταβίτ Σασόλη, αγαπητέ Σαρλ, αγαπητή Ούρσουλα, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχά, ε, θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμή ε, στου επαγγελματίε υγεία, οι οποίοι είναι εξαντλημένοι από τη μάχη κατά του COVID-19. Ε, Σα ευχαριστώ όλη η Ευρώπη και ξέρω ότι πόρο απέχουμε από τη λήξη τη μάχη. Επίση, και σε όλου αυτού που ζητούν την δύναμη τη δημοκρατία μα και την ικανότητα να αντιμετωπίσουμε δύσκολε αποφάσει, οι οποίε αλλάζουν τη ζωή εκατομμυρίων πολιτών. Θα πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη, ε, συλλογική δημιουργικότητα και καθημερινή γενοδορία. Ζούμε δύσκολες στιγμές ε, και ε, δοκιμάζει το καθένας από μας. Αλλά οι αποδείξεις και οι επιλογές που κάνουμε ε, θα τελειώσουν, αλλάξουν οριστικά τον τρόπο που ζούμε. Θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε τη ζωή μας από εδώ και πέρα από τα διδάγματα που θα αντλήσουμε από αυτή την κρίση. Έχουμε την ευθύνη λοιπόν να αντλήσουμε όλα τα διδάγματα από αυτή την υγειονομική κρίση. Δεν θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει τα πράγματα καλύτερα αν δεν είχαμε αναγνωρίσει ότι στην αρχή της κρίσης ότι ε, υπήρχαν κάποιες ε, ε, δυσκολίες και η αρχική δισταγμή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν αφήσει και αμφιβολίες στους Ευρωπαίους πολίτες. Αν θέλουμε λοιπόν να αναρώσουμε όχι μόνο από τον ιό αλλά και από τον εγωισμό μας ο οποίος ορισμένες φορές δεν μας αφήνουν να κάνουμε πράγματα. Μπορεί να φορέσουμε μάσκες για να προστατευτούμε για τον ιό αλλά θα πρέπει να πέσουν οι μάσκες και να αναγνωρίσουμε τα σφάλματά μας. Είδαμε πόσο ευάλωτα είναι τα συστήματα υγεία μα ε, και το γεγονό ότι πρέπει να έχουμε πιο εύρωστα συστήματα. Η Ευρώπη που επιθυμούμε δεν είναι αυτή των ε, ε, αχρίαστων τυχών, αλλά ελικόπτερα τα οποία θα πρέπει να διασχίζουν τα σύνορα και να πηγαίνουν τους ασθενείς εκεί όπου υπάρχουν ελεύθερες κλίνες. Η Ευρώπη που θέλουμε είναι αυτή που θα βρει ε, λύσεις για την... ασθένεια και θα μπορέσει να τις μοιραστεί. Η, ευθόρμητη συνεργασία θα πρέπει να οικοδομείται σε έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό υγεία, ο οποίο θα κάνει την ε, Ευρώπη ε, πιο αυτάρκη και πιο κυρίαρχη για την επόμενη μέρα. Για τι κρίσει αυτέ, η Ευρώπη θα πρέπει να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτέ τι κρίσει με ανεξαρτησία και θα πρέπει ευθύ εξ αρχή να σκεφτούμε αυτόν τον ευρωπαϊκό μηχανισμό υγεία, ο οποίο θα πρέπει να συσταθεί. Δεύτερον, η οικονομία. Όλοι χρησιμοποίησαμε την ίδια έκφραση, whatever it takes, ό,τι χρειαστεί. Πρέπει πλέον να περάσουμε στις πράξεις. Ε, κανένας από εμά δεν είναι σε θέση να βγει ενισχυμένος από μόνο του από αυτή την κρίση. Ε, καμία χώρα, ε, είτε ανήκει είτε δεν ανήκει στην Ευρωζώνη. Δεν θα πρέπει να είμαστε απομονωμένοι, αλλά μονιασμένοι αυτή τη φορά. Και το λέω και στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι στιγμή να παίζουμε μικρά παιχνιδάκια. Θα πρέπει να ε, δώσουμε ένα δυνατό χτύπημα με ένα νέο σχέδιο Marshall, όπως είπε η πρόεδρος Φοντερ Λάιον, και να ενισχύσουμε τα ψηφιακά θέματα και το, η πράσινη συμφωνία, το Green Deal. Θα πρέπει λοιπόν να εφαρμόσουμε αυτή τη στρατηγική αυτή τη στιγμή. Για τις επενδύσεις, ε, για την απασχόληση, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, για τις βιομηχανίες του αύριο. Η κρίση αυτή ε, δείχνει ε, και δοκιμάζει την εσωτερική αγορά η οποία θα πρέπει να αντέξει. Τρίτον, τα αυταρχικά καθεστώτα δεν είναι καλύτερα εξοπλισμένα από τις ανοιχτές δημοκρατικές κοινωνίες που βασίζονται στην ελευθερία και στη δημοκρατία για τις ε, σημαντικές αποφάσεις αναδίπλωση δεν είναι ε, ισχυρό χαρτί, είναι αδυναμία. Και με καμία κυβέρνηση η δημοκρατική Ευρώπη και τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν θα πρέπει να αμφισβητούν. Και το γνωρίζουν όλοι αυτό και ο Βίκτορ Ορμπάν. Πρέπει να κάνουμε ό,τι πρέπει, ό,τι μπορούμε για να αποκαταστήσουμε το κράτος δικαίου με όλα τα μέσα. Για όλα αυτά τα θέματα λοιπόν τίθεται το εξή ερώτημα. Ποια θα είναι η Ευρώπη μετά, ποια θα είναι η Ευρώπη μετά από αυτή την κρίση. Θα είναι ένα ε, άκαμπτο οικοδόμημα ή θα είναι ένα εύκαμπτο και ελαστικό οικοδόμημα που θα μπορεί να αντιμετωπίσει το μέλλον. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί το μέλλον μας, ε, είτε είμαστε Ρουμάνοι, Ιταλοί, ε, Δανείοι, δεν θα πρέπει να βασίζεται στην ατομικότητά μας, θα είναι ανάλογο της ε, ικανότητάς μας να συνεργαστούμε. Η κρίση αυτή αποδεικνύει και την ανάγκη να προχωρήσουμε το σχέδιο αυτό για τη μελλοντική διάσκεψη για την Ευρώπη που είναι ε, πιο απαραίτητη από ποτέ. Πρέπει να δράξουμε αυτή την ευκαιρία για να βάλουμε τάξη στον ευρωπαϊκό οίκο και με σθένος μάλιστα. Θα πρέπει να έχουμε μια πιο κοινοτική, πιο δημοκρατική Ευρώπη. Αυτή η κρίση δεν θα πρέπει να είναι ευκαιρία για να κρατήσουμε περισσότερα. Θα πρέπει να είναι μια ευκαιρία για να δώσουμε μάχη ε, κατά της ε, αυτάρκειας, κατά της υποκρισίας και των προκαταλήψεων και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη από όσα διδαχθήκαμε τα θετικά μετά αυτής της κρίσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πρόεδρε Τσόλο, Ο κύριος Καμπομενώση για την ομάδα ID. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την Πρόεδρο Φόντερ Λάιεν, τον Πρόεδρο Μισελ για την παρουσία τους και ελπίζω να είναι η τελευταία συνεδρίαση στην οποία δεν θα μπορούν να έρθουν οι συνάδελφοι στις Βρυξέλλες γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, όπως ζητούμε να εργαστούν τα εθνικά και τα περιφερικά κοινοβούλια, θα πρέπει και οι Βρυξέλλες να ε, λειτουργούν ε, απρόσκοπτα, γιατί αυτό ζητούν οι πολίτες μας. Εγώ είμαι από την περιοχή της Λιγκούρια, από τη Λομβαρδία, ε, που είναι κοντά στην πόλη μου και ο καθένας στην περιοχή μου γνωρίζει φίλους, συγγενείς που ή βρίσκονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση ή έχουν ήδη ε, χαθεί. Ίσως αυτό το οποίο δεν γνωρίζουν κάποιοι και δεν έχουν αντιληφθεί είναι την απογοήτευση όποιο αντιμετωπίζει μόνος του αυτή την κατεπίγουσα ανάγκη γιατί βρίσκεται μόνος του σε καραντίνα ή γιατί είναι μόνος του και δεν έχει την φροντίδα των ανθρώπων του και βρέθηκε στο νοσοκομείο ε, να νοσηλεύεται και αγαπητοί και συγγενείς, ε, αγαπητέ του άνθρωπα και συγγενείς που ορισμένε φορές δεν μπορούν να παραβρεθούν ότι στην κηδεία του. Ε, και φυσικά είναι και ο οικονομικός αντίκτυπος για τις επιχειρήσεις, για τους αυτοαποσχολούμενους, για τους εργαζομένους που θέλουν να επιστρέψουν στην παραγωγή και φυσικά αυτό θα είναι απαραίτητο. Θα είναι απαραίτητο να υπάρξουν κάποιες διαδικασίες ε, οι οποίες θα είναι ε, ομογενείς και συγκεκριμένες ώστε να μπορέσει το σύστημα παραγωγής να επιστρέψει με ασφάλεια, κυρίως για την ασφάλεια των εργαζομένων, να επιστρέψουμε και πάλι στην 100% παραγωγικότητα. Το πρόβλημα είναι ότι εάν εν μέρη ε, βγούμε γρήγορα από αυτή την κρίση θα είναι χάρη σε ένα σύστημα κανόνων που υπήρχαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ε, ε, για τους οποίους πρέπει υποχρεωτικά να υπάρξουν καλοί παρεκκλήσεις και είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε και κατά πόσον το σύστημα αυτό που είναι αυτό το οποίο έκανε την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια να είναι η Ήπειρος που υπήρχε η μικρότερη ανάπτυξη. Και ήταν προφανέ ότι οποιαδήποτε αιτία, σαν αυτή που ζούμε αυτή τη στιγμή, θα μπορούσε να ήταν και ένα πόλεμο ε, ή και κάποια κερδοσκοπική φούσκα όπω είχαμε πριν από κάποια χρόνια, θα υπήρξαν ακραίε δυσκολίε. Ένα σφάλμα λοιπόν που δεν πρέπει να διαπράξουμε όταν θα τελειώσει αυτή η οικονομική κρίση είναι να αναθεωρήσουμε αυτό το σύστημα κανόνων που απέτυχαν ε, σαν να μην υπήρχαν και ποτέ. Διότι συζητούμε για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που μέχρι πρώτη ήταν υπέρ τη μετεγκατάσταση μέσω εμπορικών συμφωνιών που σήμερα μας κάνουν να αντιληφθούμε ότι ε, δεν ήμασταν σε θέση να παράξουμε κάποια πράγματα. Βλέπω κάποιους προέδρους, για παράδειγμα, τον πρόεδρο της Γαλλίας που λέει ότι θα πρέπει να έχουμε πλέον ε, παραγωγική αυτονομία όχι μόνο στον τομέα της υγείας αλλά και στον τομέα της γεωργίας ε, και σε πολλούς άλλους. Η έρευνα. Πριν από λίγες ημέρες ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας παρετήθηκε καταγγέλλοντας ε, την αδυναμία να εργαστεί στον τομέα αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όλοι χρησιμοποιούν τον όρο αλήθεια, κατάχρηση του όρου γίνεται και προσπαθούμε να δώσουμε μια ευρωπαϊκή προοπτική ε, προσπαθώντας να δώσουμε μια προοπτική που κατά την άποψή μου είναι αποκλειστικά και μόνον αυτή της επικοινωνία που έχει στόχο να προστατεύσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι θύμα του εαυτού τους, ε, του τρόπου με τον οποίο επικοινώνησε τα τελευταία χρόνια. Πλασαρίστηκε στους πολίτες ως ένα σύστημα το οποίο δεν είναι στην πραγματικότητα με ένα προπολογισμό ο ίσως θα μπορούσε μπορούσε να είναι χρήσιμο, θα το επεξεργαστούμε αυτό, αλλά τελικά θα δώσει πενιχρούς πόρου. Αυτό που χρειάζεται πρωτίστω είναι οι πολίτες να είναι ελεύθεροι, ε, οι χώρες να είναι ελεύθερες να κάνουν την πολιτική του να έχουμε ένα σύστημα ε, που δεν είναι αυτό του Federal Reserve ή της Τράπεζας της Αγγλίας και φυσικά θα πληρώσουμε τι συνέπειε. Να μην μιλήσω για το γεγονό ότι εντό ολίγου θα έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο οποίο ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού, ο, ο, θα πάει χωρί εντολή διότι υπάρχουν και έρηδες και μία συζήτηση για το μηχανισμό σταθερότητας, ε, το EMS, ε, το οποίο ε, οδήγησε σε πολύ μεγάλο διχασμό. Εγώ είμαι βέβαιος ότι η Ιταλία θα τα καταφέρει. Δεν είμαι βέβαιος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να ξεπεράσει αυτή την κρίση. Η Ευρώπη και τα κράτη-μέλη και η Ιταλία θα τα καταφέρουν, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το πιστεύω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Φίλοι, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συμπολίτε, απευθύνομαι σε εσά από το ημικύκλιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, εκεί όπου χτυπάει η καρδιά της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας κανονικά. Σήμερα αυτή η καρδιά χτυπά πιο αργά. Όλοι έχουμε επηρεαστεί από την πανδημία. Οι μέρες αυτές ε, είναι θλιβερές. Δεν μπορούμε παρά να σκεφτούμε τις δεκάδες χιλιάδες θύματα, τους συγγενείς τους, ε, τις δυσκολίες που είχαν ε, οι συγγενείς ε, να θρηνήσουν τους αγαπητούς τους και θέλουμε να αναγνωρίσουμε όλους εκείνους που καθημερινά προσφέρουν υπηρεσίες με κίνδυνο της υγείας τους στους ασθενείς και στα θύματα. Έχουμε στην καρδιά μας επίσης εκείνους που παρά την πανδημία βρίσκονται στις θέσεις εργασίας του ώστε οι κοινωνίες μας να συνεχίσουν να ζουν πολύ απλά. Η Ευρώπη δεν έχει αντιμετωπίσει τέτοια κρίση από το 1945 και μετά. Το σοκ που δημιούργησε ο κορονοϊός δείχνει τα ελαττώματα των κοινωνιών μας. Ε, πράγματα που πολλοί πολιτικοί μέχρι σήμερα δεν ήθελαν ούτε να ακούν ούτε να βλέπουν. Πολλοί ανακαλύπτουν ξαφνικά ότι η λιτότητα σκοτώνει όταν βλέπουμε πόσοι άνθρωποι μεγάλη ηλικία πεθαίνουν. Μα δείχνει πω η παγκοσμιοποίηση που καθοδηγείται μόνο από το κέρδο αποδυνάμωσε τις κοινωνίες μα. Βλέπουμε τις καταστροφές ε, που δημιουργήσαν ε, οι κοινωνικές ανισότητες. Εκατομμύρια Ευρωπαίοι πέρασαν μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα σε αναγκαστική ανεργία. Πολλοί δεν έχουν χρήματα για να τραφούν. λόγω της ανεπάρκειας των κυβερνήσεών μας, ε, πόσα καταστήματα χρειάστηκαν να κλείσουν. Πράγματα, ε, άνθρωποι που μέχρι ε, σήμερα ήταν στατιστικά στοιχεία ότι βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας, ξαφνικά δεν έχουν να φάνε. Η κοινωνική προστασία δεν είναι επαρκής και όπως φαίνεται ξαφνικά η αβεβαιότητα υπάρχει παντού, σε όλη την Ευρώπη σήμερα. Σήμερα αυτοί οι αόρατοι άνθρωποι δεν μπορούν πια να, να τους ξεχνάμε. Στο πλαίσιο αυτής της πανδημίας εγώ ανησυχώ, διότι θα έχει σοβαρές συνέπειες στις κοινωνίες μας πρώτος κίνδυνος. Για άλλη μια φορά, οι πιο αδύναμοι θα είναι αυτοί που θα πληρώσουν ε, τα σπασμένα μια κρίσης για την οποία δεν έχουν ευθύνη. Σκέφτομαι εκείνους που είναι ε, χωρίς ε, κατοικία, ε, που η θέση εργασία του κρέμεται από μια κλωστή. Ε, Αυτού που περιμένουν υπό απάνθρωπε συνθήκε να μπουν στην Ένωση, στου καταβλισμού ε, προσφύγων, που προσπαθούν να φύγουν από χώρε που υποφέρουν από πόλεμο και από την κλιματική αλλαγή και ξαφνικά πλήττονται από την πανδημία. Αν αντιμετωπίσουμε τα πράγματα όπως πριν από 10 χρόνια στην οικονομική κρίση, θα διαραγούν οι δεσμοί των κοινωνιών μας και θα θέσουν σε κίνδυνο την ύπαρξή μας. Δεύτερος κίνδυνος, οι δημοκρατίες μας μπορεί να αποδυναμωθούν σημαντικά, όπως στην Πολωνία για παράδειγμα, ή να ανασταλούν τελείως όπως στην Ουγγαρία. Ξαφνικά ε, οι πρόεδροι να αναλάβουν ε, όλα τα ενία ε, εις βάρος του ανεξαρτητού τύπου και των κοινοβουλίων και να περάσουν σε κράτη μόνιμης παρακολούθησης. Τρίτος κίνδυνος, η πενδημία να αποτελέσει ένα τέλειο άλοθη για να εκμεταλλευτούν κάποιοι α, χωρίς όρια τα πάντα στον πλανήτη μας ώστε να εκμεταλλευτούν ε, αυτό προσπαθούμε εμείς να κάνουμε να συνεχίσουν να ζουν οι κοινωνίες μας σωστά η κλιματική απορρίθμιση, η βιοπικιλότητα, οι πόροι που εξαντλούνται δεν σταματούν από τον κορονοϊό. Το να επανακινήσουμε τον διεθνή μηχανισμό χωρίς προγραμματισμό μπορεί να μας οδηγήσει σε καταστροφή, σε μεγαλύτερη καταστροφή των κοινωνιών μας από ότι η πανδημία. Τέταρτος κίνδυνο, η κρίση αυτή να σκοτώσει την διεθνική δημοκρατία, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Όταν η πανδημία έφτασε στις ακτέ μας, πολλά κράτη-μέλη δεν θέλησαν να στείλουν εξοπλισμό σε άλλα κράτη που τον είχαν ανάγκη και αυτό ήταν ε, το κέριο πλήγμα. Και σήμερα θα χρειαζόμαστε μια συνολική στρατηγική για να ανταποκριθούμε στην ε, πανδημία και για να εικονοδίσουμε τις κοινωνίες μας. Εμείς είμαστε πεπισμένοι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τα μέσα συλλογικά για την ανοικοδόμηση της οικονομίας της, εφόσον φυσικά κινητοποιηθούμε όλοι μαζί. Και αν είναι να χρεωθούμε, θα πρέπει να χρεωθούμε μαζί για να εξοφλήσουμε μαζί. Το να αφήσουμε κάθε χρόνο, κάθε κρατό μέλο μόνο του, σημαίνει ότι καταδικάζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Νομισματική Ένωση. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να απευθυνθώ ε, στον κύριο ε, Βούστρα, τον ε, Υπουργό Οικονομικών τη Ολλανδία και όλου όσου τον υποστηρίζουν. Και θέλω να του πω ότι η χώρα του, όπω η Γερμανία και η Φιλανδία και η Αυστρία και όλε αυτέ οι χώρε που θεωρείται ότι είναι υγιεί, ήταν οι πρώτε που ε, επωφελήθηκαν οικονομικά από την ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Και του λέω δυνατά, η κοινωνική και οικονομική αλληλεγγύη είναι το τίμημα που πρέπει να πληρώσετε για όλα αυτά τα ωφέλη. Και είναι σκανδαλώδες το ότι ακούμε ξαφνικά από Ολλανδούς πολιτικούς μαθήματα περί δημοσιονομικής πειθαρχίας, ενώ αυτοί εδώ και δεκαετίες στερούν τα άλλα κράτη-μέλη από φορολογικά έσοδα τα οποία δικαιούνται. Αγαπητοί συμπολίτε, σε αυτή τη ε, φάση η εικόνα που σα δίνω μπορεί να φαίνεται σκοτεινή, αλλά ξέρετε, ε, εμά ε, οι πράσινοι, οι πειρατέ δεν είμαστε αυτοί που τα παρατάμε όταν μένεται η καταιγίδα. Το χειρότερο είναι βέβαιο μόνο αν υποταχθούμε σε αυτό όλη αυτή η κρίση μπορεί να ανοίξει νέους οριζόντες για τις κοινωνίες μας και να μας δώσει ευκαιρίες απρόσμενες. Για παράδειγμα αυτή η ιεραρχία ε, των ε, θέσεων εργασίας ε, όπου στην κορυφή βρίσκονται τα αφεντικά, οι traders, ε, οι επενδυτές ε, και οι ποδοσφαιρικοί στάρα. Σήμερα ξαφνικά ανακαλύπτουμε πόσο αναγκαίοι είναι άλλοι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που μας φροντίζουν στα νοσοκομεία, που καλλιεργούν τη γη, τη γη που παράγουν τα τροφιμά μας, ε, που μας βοηθούν να μετακινούμαστε, που μαζεύουν τα σκουπίδια μας. Αυτοί που χθε και σήμερα και αύριο μας μαθαίνουν πράγματα που μας διευρύνουν τους οριζοντές μας δεύτερο θύμα της πανδημίας είναι η ιδέα, ότι ε, η αγορά είναι αυτή στην οποία βασίζεται ολόκληρος ο πλανήτης. Αυτό η ιδεολογία όπως φαίνεται δεν θα διατηρηθεί. Ε, αυτή η περάσπιση του γενικού συμφέροντος ξεκινά από τη ζωή και από τους δημοκρατικούς θεσμούς και τις δημόσιες υπηρεσίες που οργανώνονται για προς όφελος όλων. Ο κορονοϊός μπορεί να πλήξει μοιραία τον άνθρωπο ως αρχηγό της φύσης. Η φύση είναι κομμάτι μας. Από αυτήν εξαρτόμαστε για να ζούμε. Για να είμαστε σωστοί και οι θα πρέπει να τηρούμε τους κανόνες. Ένα άλλο θύμα του ιού μπορεί να είναι αυτή η αιμονή, να έχουμε όλο και περισσότερα, πιο γρήγορα, πιο μεγάλα, πιο μακριά. Κάτι που μας ε, οδηγεί στο να ασκούμε πίεση μονίμως σε όλο τον πλανήτη. Διότι ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι η παγκόσμια κλίμακα δεν είναι πάντα η καταλληλότερη. Το να μεγιστοποιούμε την αποτελεσματικότητα τόσο υπερβολικά δυνάμει του κέρδους γίνεται πάντα εις βάρος της ε, αντοχής μας να αντέξουμε σοκ και να ανταποκριθούμε σε αυτά. ο όμο οικονομικός, ο οικονομικός άνθρωπος μπορεί τελικά να χάσει μέσα από όλα αυτά προσπαθώντας να μεγιστοποιεί το κέρδος του διότι ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι η ζωή σίγουρα υπάρχει, ναι, με οικονομική και ηλική άνεση, αλλά χρειάζεται και χρόνο, χώρο, ιδέες που μας επιτρέπουν να σχετιζόμαστε με τους άλλους και με τον κόσμο. Αγαπητοί συμπολίτες, η πανδημία ξαφνικά ανακόπτει όλο τον πλανήτη, την ανθρωπότητα και πρέπει να την εκμεταλλευτούμε για να επιλέξουμε μαζί τι δρόμο θα ακολουθήσουμε εμείς και οι κοινωνίες μας. Για μας είναι αδιανόητο και εντελώς ανεύθυνο να θέλουμε απλά να επανεκκινήσουμε το μηχανισμό ε, εκεί που βρισκόμασταν πριν τον κορονοϊό. Ας ε, ε, μην υιοθετήσουμε απλουστικές λύσεις. Η πανδημία λόγω του φιλελευθερισμού μας οδήγησε σε τεράστια προβλήματα. Ωστόσο, η αυτάρκεια και το να αντιπλανόμαστε στον εαυτό μας δεν αποτελεί εγγύηση. Μεταξύ του παγκοσμίου και του τοπικού θα πρέπει να δημιουργήσουμε νέες ισορροπίες βάσει των διαφορετικών πλούτων των χωρών μας. Τι καλούμαστε να κάνουμε, να ανασχεδιάσουμε τον τρόπο λειτουργία των κοινωνιών μα, με πηξίδα τη ζωή, μία ζωή αξιοπρεπή για όλου και όλε. και όχι το κέρδος αυτό απαιτεί ευφυΐα, δημιουργικότητα, συλλογική. Πέραν της άμεσης ε, καταπολέμησης της πανδημίας θα πρέπει να προετοιμάσουμε αυτή την κινητοποίηση με όλους όσους σήμερα ε, ήδη υποστηρίζουν νέους τρόπους ζωής, ε, μετακίνησης, διαβίωσης. Είμαστε έτοιμοι. Για να κλείσω, θέλω να πω καθαρά, εντός των ευρωπαϊκών θεσμών και ειδικότερα απευθυνόμενο στους αρχικού κρατών και κυβερνήσεων που εκπροσωπεί εδώ ο πρόεδρος του Συμβουλίου που θα συνεδριάσετε πάλι την επόμενη εβδομάδα δεδομένη τη πανδημία και των συνεπειών τη, ο λόγο ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διακυβεύεται. Αν δεν καταφέρουμε να δράσουμε αλληλέγγυα μπροστά σε αυτή την πρόκληση που μας πλήττει όλους, τι νόημα έχει η ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για μας είναι σαφές ότι οι εθνικοί εγωισμοί θα μας οδηγήσουν στο να αναβαγίσουμε. Μαζί θα πρέπει να βρούμε το δρόμο για το μέλλον μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Πρόεδρε Λάμπερτ. Πάμε στην απομακρυσμένη, σε μια απομακρυσμένη σύνδεση. Πρόεδρε Φίτο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας όλοι. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε αυτή την ευκαιρία. Εύχομαι και εγώ να μπορέσουμε να επανέλθουμε γρήγορα στις εργασίες μας εντός της αίθουσα της Ολομέλειας. Και εγώ ήθελα να εκφράσω τη συμπαραστασή μου ως Ιταλός ε, στους πολυάριθμους ε, ανθρώπους που έψαν θύματα δυστυχώς ε, καθημερινά μαθαίνουμε για αυτούς λόγω αυτής της δραματικής κατάστασης που αντιμετωπίζουμε. Και εγώ θα ήθελα να υπογραμμίσω πόσο άριστο είναι το έργο που προσφέρουν ε, το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό, οι εθελοντές, οι δυνάμεις της τάξης, ε, οι, δυνάμεις, οι στρατιωτικές δυνάμεις που βοηθούν να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δραματική πανδημία. Θεωρώ ωστόσο ότι είναι απαραίτητο αυτή τη στιγμή να μην ε, εκφράζουμε μόνο τι φοβόμαστε ότι θα συμβεί, αλλά να ξεκαθαρίσουμε λίγο και το τι συνέβη. Και πρέπει να πούμε πολύ σαφώς ότι η Ευρώπη ήταν εντελώς απροετοίμαστη για αυτό το ρόλο συντονισμού που χρειάστηκε να διαδραματίσει. Κάποια κράτη μάλιστα ε, έδειξαν ε, ε, σοβαρά εγωιστική στάση σε στιγμή που η λέξη αυτή η αλληλεγγύη που τόσο συχνά ακούμε έπρεπε να υλοποιηθεί και σήμερα το πρωί έπρεπε να είναι στο επίκεντρο κάποιες χώρες ε, ε, έπρεπε να συμπαρασταθούν στα θύματα της πανδημίας αυτής. Αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε προσεκτικά και βάσει των όσων θα γίνουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες και ημέρες και τους μήνες διότι δεδομένης αυτής της υγειονομικής ε, τραγωδίας ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε να προβληματιστούμε σοβαρά για το τι θα πρέπει να υλοποιήσει οικονομικά η Ευρώπη ώστε αυτή η τραγωδία να μην μετατραπεί σε οικονομική τραγωδία και να καταστρέψει οδηγώντας μας σε μια αναπότρεπτη κρίση στην Ευρώπη και στα κράτη-μέλη. Οπότε και εδώ θα πρέπει να κάνουμε κάποιες ε, δηλώσεις αναγκαίες. Πρώτον, υπάρχει μια δυσάρεστη αίσθηση ότι συνεχίζουμε να μιλάμε όπως μιλούσαμε πριν ε, δύο μήνες, πριν από αυτή την πανδημία, τόσο όσον αφορά τις προθεσμίες για τις συζητήσεις, ε, τις διαπραγματεύσεις και τις αναστολές, αλλά και για κάποιες στάσεις που το ψήφισμα που θα ψηφίσουμε σήμερα μάλιστα αναδεικνύει και που η ομάδα μας καταγγέλει στεναρά θα πρέπει να βρεθεί χρόνος ε, και ε, χρόνος και χώρος ε, για διάφορες διαπραγματεύσεις για το άρθρο 7 κατά των κυβερνήσεων της Πολωνίας και της Ουγγαρίας. Εμείς θεωρούμε ότι είναι ανεπίτρεπτο δεδομένη της κατάστασης που έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στις λύσεις οικονομικού χαρακτήρα οι οποίες θα πρέπει να δοθούν καθαρά να είναι συγκεκριμένε και αποτελεσματικές, ούτω ώστε να δώσουμε απαντήσεις στους πολίτες, στους εργαζομένους, στι επιχειρήσεις μας, σε τομείς που έχουν πληγεί σημαντικά, όπως ο τουρισμός, οι μεταφορέ, η γεωργία, η μεταποίηση, οι τομείς ε, που βρίσκονται σε δραματική κατάσταση και χρειάζονται σαφή μέτρα που θεωρούν ότι οι ευρωπαϊκές απαντήσεις, ε, τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Αυτές οι πρώτες πρωτοβουλίες ναι μεν τους βοηθούν αλλά ε, χαρακτηρίζονται από γραφειοκρατία, από πολλά γραφειοκρατικά εμπόδια. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πιο ευρέω από ό,τι απλά σε θέματα ευρωπαϊκού προπολογισμού. Κάποιοι υπερασπίζονται ακόμα σαφώ κάποια σημεία που έχουμε συζητήσει του τελευταίου μήνε. Ο προπολογισμό πρέπει να τροποποιηθεί σημαντικά αλλιώ. Είναι αδιανόητο να μπορούμε να συζητάμε τα προγράμματα που είχαν αποφασιστεί πριν την κρίση αυτή, το Green Deal. Στο πλαίσιο που ζούμε σήμερα πρέπει να ανασχεδιάσουμε τις επιλογές που θα χρησιμοποιήσουμε για το μέλλον. Και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι απαραίτητο να δώσουμε και απαντήσεις σαφείς και αποτελεσματικές με εργαλεία καινοτόμα τα οποία θα δείχνουν ότι η Ευρώπη είναι πραγματικά αλληλέγγυα. Εγώ θεωρώ ότι αυτό αναμένουν από εμάς οι Ευρωπαίοι πολίτες και έτσι θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε εμείς ως συντηρητική σε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστούμε κύριε Φίτο. Κύριε Όμπρη έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, στο όνομα της ομάδας της Ευρωπαϊκής Αριστεράς δεν μπορώ παρά να συμμεριστώ τις σκέψεις των λοιπόν ομιλητών ε, που πάνε βεβαίως στα θύματα, ε, στο ιατρικό προσωπικό, η έκκληση ε, αλληλεγγύη απέναντι στην υγειονομική αλλά και οικονομική κοινωνική κρίση που χτυπάει την Ευρώπη. Θα πρέπει να υπάρξει μια συλλογική ε, προσπάθεια χωρίς και πέρα από συμφέροντα. Είναι απαραίτητο ένα σύστημα υγείας να προστατεύει όλους. Όμως, να τα πούμε τα πράγματα σωστά, ευθύς εξ αρχής. Όλα αυτά τα λόγια δεν έχουν κανένα νόημα όσο απλά θα παρακολουθούμε το τι συμβαίνει. Πρέπει να πάμε πέρα από αυτό. Πρέπει καταρχήν να καταλάβουμε γιατί συμβαίνει αυτή η καταστροφή. Πώ μπορούμε να εξηγήσουμε ότι σε αυτό το κοινό ψήφισμα που μα υποβάλλεται δεν λέγεται ούτε μία λέξη, ούτε μία αναφορά στην ευθύνη που φέρουν οι, δημοσιονομικέ περικοπέ για το πώ είναι τα υγειονομικά μα συστήματα σήμερα. Είναι ο απολογισμός της λιτότητας καταστροφικός. 120.000 ε, κρεβάτια τα οποία χάθηκαν στη Γαλλία, 14% των δυνατότητών μας. Ε, ναι, κύριε και κύριοι, η λιτότητα σκοτώνει. Δεν μπορούμε εμείς να κλείνουμε τα μάτια απέναντι στο γεγονός αυτό. από το 2011 έως το 2018 63 φορές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τα κράτη-μέλη να μειώσουν τις γερμανικές δαπάνες. Τα φιλελεύθερα, οι φιλελεύθερες κυβερνήσεις βέβαια αυτό το πρόσχημα περίμεναν, αυτό το άλοθη για να καταστρέψουν τα, τα δημόσια νοσοκομεία. Και τώρα αντλούμε πολιτικά συμπεράσματα. Είναι καθήκον μας να αρνηθούμε οποιαδήποτε προϋπόθεση λιτότητας για να μπορέσει κάποιος να χαίρει ε, ε, προγραμμάτων ενίσχυσης όπως ο μηχανισμός αλληλεγγύης. Η Ιταλία ενώ ο λαός της πεθαίνει δεν ξέρει αν πρέπει να δεχτεί αυτό το δηλητηριασμένο δώρο της Ένωσης και πραγματικά εγώ ντρέπομαι που σιωπούμε απέναντι σε αυτά τα διλήμματα τα οποία επιβάλλουμε στους Ιταλούς ότι ή πρέπει να υποκύψουν ή να πεθάνουν αυτή η κατάσταση με το δημόσιο χρέος το οποίο χρησιμοποιεί το δαμόκλειος σπάθη πάνω από τις κυβερνήσεις πρέπει να σταματήσει και βεβαίως ε, βλέπουμε τι λένε οι εργοδότες, τι λένε οι κυβερνήσεις. Η κρίση κοστίζει ακριβά. Θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες. Θα πρέπει να εργαστούμε περισσότερο. Ειλικρινά, ε, δεν χρειάζεται να τα ακούσουμε ε, για άλλη μια φορά. Τα έχουμε ακούσει πολλές φορές την κρίση θα την πληρώσει ο λαός. Ιδίως αυτοί οι οποίοι είναι οι πιο φτωχοί και την πληρώνουν ήδη. Όλα αυτά που λέτε λοιπόν ακούγονται λίγο κούφια όταν ζητάτε νέες θυσίες. Όταν λέμε ότι η μόνη λύση ουσιαστικά είναι η λιτότητα. Λες και αυτό το χρέος είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε ποτέ. Μα ζητάτε να σφίξουμε το ζωνάρι για ακόμα μερικές δεκαετίες δεν πρέπει να μείνουμε φυλακισμένοι σε αυτή τη λογική. Θα πρέπει να θυμηθούμε τι έλεγε ο φυλακισμένος του Αλμπέρ Καμού. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να ξεφύγω από το μηχανισμό του να ξέρω κατά πόσο το αναπόφευκτο μπορεί να οδηγήσει κάπου. Αυτή, το που οδηγεί αυτό γνωρίζουμε ποιο είναι. Ζητούμε να υπάρξει δίκαιη κατανομή της κρίσης αυτής, να πληρώσουν οι πλούσιοι, το μεγάλο κεφάλαιο. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η νομισματική πολιτική για να μην πάμε προς τη λιτότητα. Γιατί οποιαδήποτε ε, κοινή προσέγγιση του χρέους ε, δεν γίνεται δεκτή. Γιατί να μην επενδύουν, ε, για να μην χρηματοδοτεί άμεσα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα τα κράτη-μέλη όπως κάνει η Τράπεζα της Αγγλίας. Γιατί να μην διαγράψουμε προοδευτικά το χρέος ε, των χωρών όπως έχει γίνει και στο παρελθόν. Ήρθε η στιγμή όλα αυτά τα ταμπού να τα συντρίψουμε. Είναι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση σήμερα, αλλά και την κλιματική πρόκληση του μέλλοντος. Όλα αυτά τα διακευόμενα όμως, δυστυχώς, εσείς τα αγνοείτε. Ένα ισχυρό κοινοβούλιο αυτό θα πρέπει να περασπιστεί για να μπορέσει να επηρεάσει τη συζήτηση. Συζήτηση από την οποία συχνά βρίσκεται απ' έξω. Δεν πρέπει να είμαστε απλά θεατές βουβοί θα πρέπει αυτά τα παλιά δόγματα τα οποία μας οδηγούν στην καταστροφή να τα παραμερίσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ομπρί. Ακολουθεί Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Φοντελάγεν και τον κύριο Μισελ για την παρουσία τους εδώ ε, και για τον ε, ηγετικό ρόλο που έχουν παίξει στην αντιμετώπιση αυτή τη κρίση. Όμω, στι στιγμέ τη κρίση αντιλαμβανόμαστε πόσο περιορισμένο είναι το πεδίο δράση των οργάνων μα. Αναφερθήκατε στο ζήτημα του μέλλοντο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφερθήκατε σε αυτό το μέλλον το οποίο εξαρτάται από το πώ θα διαχειριστούμε αυτή την κρίση. Δυστυχώ, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ένα πολύ καλό παρελθόν στην αντιμετώπιση και διαχείριση κρίσεων. Η κρίση του 2008, η χρηματοοικονομική κρίση, έχει ακόμα επιπτώσεις και η Ευρώπη εκεί απέτυχε. Οι επιπτώσεις είναι απίστευτες και είναι καταστροφικές ιδιαίτερα στην περιφέρεια της Ευρωζώνης. Το θέμα της μετανάστευσης επίσης έτυχε λαθασμένης διαχείρισης. Καταστροφική διαχείριση και βεβαίως και εδώ οι επιπτώσεις μας ακολουθούν ακόμα και σήμερα. μπορούμε μόνο να ελπίζουμε ότι η διαχείριση της κρίσης του κορονοϊού θα είναι διαφορετική. Κύριε Μισελ, αναφερθήκατε στην πίεση που προέρχεται από τους πολίτες για να μεταρρυθμίσουμε τους θεσμούς μας. Έχετε δίκιο. Ε, η μεταρρύθμιση των ε, θεσμών είναι απαραίτητη με βάση την κρίση αυτή. Διότι εάν δεν έχουμε μεταρρύθμιση, οι Ευρωπαίοι πολίτες θα ξεγράψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα κινηθούν προς λύσεις που φαίνονται πιο σαφείς, πιο αποτελεσματικές. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μάθει και δεν προσαρμοστεί, οι εχθροί της πολύ γρήγορα θα δακτυλοδείξουν τα προβλήματά της και θα κεφαλοποιήσουν τα ωφέλη. Μιλήσαμε πολύ για αλληλεγγύη, αλληλεγγύη και επικουρικότητα. Θα πρέπει τα ζητήματα να επιλύονται τοπικά όταν γίνεται. Και υπάρχουν βεβαίω ε, ζητήματα που μπορεί να είμαστε πιο αποτελεσματικοί σε εθνικό επίπεδο. Όμω οι περισσότερε προκλήσει που αντιμετωπίζουμε χρήζουν διασυνορική συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο, ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θεσμική λοιπόν μεταρρύθμιση απαραίτητη και ό,τι κάνουμε σήμερα θα πρέπει να μα προετοιμάσει για το μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Κύριε Γκενγκεσί, ακολουθεί η κυρία Ντελάγκη για δύο λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Την περσμένη φορά που μίλησα εδώ, αναφέρθηκα στους πραγματικούς ήρωες αυτής της κρίσης, όπως ε, η αδερφή μου, που είναι ορθοπαιδικός, ε, που συνήθως ε, διορθώνει γόνατα, αλλά πλέον εργάζεται στο Μάρσιξ στο νοσοκομείο αντιμετωπίζοντα τον κορονοϊό και είδε με τα μάτια της τι κάνει αυτός ο καταστροφικός ιός. Άνθρωποι οι οποίοι μένουν μόνοι τους και πεθαίνουν μόνοι τους, δεν έχουν συγγενείς πρόσβαση σε αυτούς και γιατροί οι οποίοι έχουν μάθει να θεραπεύουν, να χάνουν την υπομονή τους. Ε, πραγματικά, ε, βεβαίως το Συμβούλιο αποχώρησε από τη συζήτηση. Θέλω να πω όμως στο Συμβούλιο ότι εδώ δεν χρειάζεται μια θεωρητική γραφειοκρατική συζήτηση για την ενιαία αγορά Βεβαίω και η ενιαία αγορά είναι στην καρδιά τη Ευρωπαϊκή ανάκαμψη ε, σε οικονομικό πεδίο που θα ακολουθήσει και βεβαίω οι επενδύσει είναι πολύ σημαντικέ ε, Η χρησιμοποίηση του προπολογισμού μα ω ένα πραγματικό εργαλείο αλληλεγγύη. Όμω αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι μάσκε. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι προστατευτικό υλικό. Χρειαζόμαστε μια Ευρώπη με καρδιά που δείχνει ότι μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Ότι ποτέ δεν πρόκειται να είμαστε εξαρτημένοι από άλλους όπως είμαστε τώρα σε ό,τι αφορά το ιατρικό μας εξοπλισμό, σε ό,τι αφορά τα φάρμακα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι αλληλεγγύη ενδράση και αναφέρομαι στα άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν από την Ολλανδία στη Γερμανία παραδείγματος ε, χάριν. Δεν χρειαζόμαστε ε, να ακούμε ε, αυτούς που λένε ότι η Ρωσία ενισχύει περισσότερο την Ιταλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί αυτό δεν είναι αλήθεια. Και αυτό που τέλος χρειαζόμαστε είναι μια Ευρώπη που θα μάθει από τα λάθη της. Έγιναν λάθη όταν πάρθηκαν τα πρώτα μέτρα για τον κορονοϊό. Άλλα έκανε το ένα κράτος μέλος, άλλα έκανε το γειτονικό κράτος μέλος. Και το Συμβούλιο θα επαναλάβει το ίδιο λάθος. Η Κομισιόν θέλει να προτείνει ενότητα σε ό,τι αφορά την εξόδου και τα κράτη-μέλη θέλουν να τη σταματήσουν. Και λέω στην Κομισιόν, πολύ καλώς έχετε προετοιμάσει κάποιε γραμμές. Πρέπει να δείξετε ε, στεναρότητα και να δείξετε στην αδερφή μου και σε όλους τους άλλους ότι μπορείτε να φέρετε αποτέλεσμα και να βελτιωθείτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Ντελάνγκε. Ακολουθεί ο κύριος Μπενιφέη για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ευπρόσδεκτα τα μέτρα τα οποία λήφθησαν μέχρι τώρα για τον κορονοϊό, αλλά θα πρέπει να αυξηθεί το επίπεδο φιλοδοξία και να υπάρχουν απτά ωφέλη για όλου του πολίτε, ιδίω για τι πιο ευπαθείς ομάδε αυτή τη κρίση. Ε, Αυτόχθονε, γυναίκε, ε, άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένου. Ε, είδαμε τι τροπολογίε για τη ΦΕΑ, το Ταμείο για τι πιο ευπαθείς ομάδε, που θα χρειαστεί περισσότερου πόρου στον επόμενο προπολογισμό. Οι εκτιμήσει του Διεθνού Νομισματικού Τομείου προβλέπουν κατάρρευση του ΑΕΠ ε, κατά 7,5 ποσοστίας μονάδε. Επομένω, είναι πάρα πολύ σημαντικό το έκτακτο σχέδιο τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεω ή το ταμείο το οποίο προβλέπεται από το μέσο ΣΟΥΛ για να υποστηρίξουμε το εισόδημα και την θέσει εργασία. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα τεράστιο οικονομικό σχέδιο ανάκαμψη. Συζητήθηκε το να χρησιμοποιηθεί τα 410 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Σταθερότητα ε, χωρί ε, όρου. Κάθε χώρα θα αξιολογήσει αν θα το χρησιμοποιήσει αλλά θεωρούμε ότι αυτό δεν επαρκεί σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό ακριβώ και είμαι περίφερο που σήμερα το Κοινοβούλιο υποβάλλει ένα ψήφισμα το οποίο θέτει επιτάπητο ε, τα ε, ομόλογα ανάκαμψη ω μέσο για να μπορέσουμε να καλύψουμε τι κοινέ υποχρεώσει σε κοινοτικό επίπεδο, κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχωρήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Απριλίου. Δεν είναι απλώ για μία ε, ad hoc ε, βοήθεια προ τι χώρε, αλλά θέλουμε να διατηρήσουμε τι επόμενε γενναίε και το κοινωνικό ιστό. Η πρόεδρο Φοντερλάν σήμερα αναφέρθηκε στον Αλτιέρο ε, Σπιρλόινιλι και στο Βεντοτένελα. Θα πρέπει να σταθούμε στο ύψο αυτή τη ε, ιστορία, όχι να την αναφέρουμε απλώ. Δεν το λέω μόνο για την πρόεδρο αλλά για όλου του ηγέτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει να χάσουμε χρόνο, δεν έχουμε ε, χρόνο. Η μεγάλη πλειονότητα των ε, Ευρωπαίων μα ζητούν να είμαστε στο ύψο τη πρόκληση και εγώ πιστεύω ότι έχουν δίκιο. Α μην του απογοητεύσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μπενιφάη. Ο ε, Σεζούνε, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να πιστέψω ότι το κείμενο που θα ψηφίσουμε σήμερα είναι το πιο σημαντικό του ενήλικου βίου μου. Γιατί αυτό, γιατί πιστεύω ότι αυτό το ψήφισμα απορρέει από τον ευρωπαϊκό λαό. Σε αυτή τη φρικτή κρίση που καταφέραμε μέσω αυτού του κειμένου να βρούμε το ευρωπαϊκό γενικό συμφέρον δεν είναι ε, κάτι το οποίο είναι απλώς για την τη Δύση, δεν είναι ιδιοκτησία κανενός, καμίας πολιτικής οικογένειας, είναι απλώς ε, για τους ε, ανθρώπους του οποίου φροντίζουμε στο Βέργαμο, στην ε, Μαδρίτη και που ζητήσαμε μια εξαιρετική υγειονομική στρατηγική για τους ταμείες, για τους οδηγούς λεωφορείων, τις οικογένειες που θέλουμε πραγματικά να έχουν μια κυρίαρχη Ευρώπη για να παράγουν μάσκες και προστατευτικό εξοπλισμό. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τι μικρέ επιχειρήσει που ζητούν περισσότερα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Είναι για του δημοκράτε αυτή τη Υπέηρου, τους οποίου ε, ε, ε, υπερασπίζονται το κράτο δικαίου στην Ουγγαρία. Και τέλο για τα παιδιά μα. είτε από τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Σλοβακία, την Ολλανδία και όποιον θέλει να μπει στην αγορά εργασία στα επόμενα 3-5 χρόνια και θέλουμε να του προστατεύσουμε και θέλουμε να επενδύσουμε από κοινού. Να επενδύσουμε από κοινού αναλαμβάνοντας ε, από κοινού το χρέος χωρίς ε, ε, ε ομολογοποίηση των προηγούμενων χρεών ε, και αμοιβεοποίηση των προηγούμενων χρεών και θα πρέπει να το κάνουμε όλοι μαζί. Και φυσικά ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντα προσπαθεί να λάβει υπόψη τι ε, φιλοδοξίε και τι ελπίδε των ευρωπαϊκών λαών. Εκπροσωπούμε διάφορε πολιτικέ ομάδε από όλη την Ευρώπη. Είμαστε ο ευρωπαϊκό λαό ε, που ε, εκλεγόμαστε από του Ευρωπαίου και καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Υπάρχει συμφωνία. δεν θέλω φυσικά να προδικάσω το αποτέλεσμα τη ψηφοφορία, αλλά καταλήξαμε σε συμφωνία. Πώς γίνεται λοιπόν σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση να φαίνεται τόσο διχασμένη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, αναφέρεται σε μια ευρωπαϊκή κοινή γνώμη ε, που συμφωνεί σε πολύ μεγάλο βαθμό με το δικό μα το ψήφισμα. Πώς, γιατί δεν το λαμβάνει υπόψη. Και θα ήθελα να δώσω μια συμβουλή στο Συμβούλιο. Κύριε Αρχηγή Κρατών και Κυβερνήσεων, προσπαθείτε να καταλήξετε σε μια συμφωνία, δεν χρειάζεται να ψάχνετε παραπέρα. Να, τι, εδώ η συμφωνία. Περιλαμβάνει όλες τις φιλοδοξίες και είναι η έκφραση του ευρωπαϊκού λαού, η αποτελεσματικότητα, η δημοκρατία, οι αξίες μας. Επομένως, ε, τίνεται δίκο νους στο Κοινοβούλιο, στους πολίτες, στους ευρωβουλευτές δεν συμπεριφερθήκαμε εμείς εδώ ως ε, αρχηγοί κομμάτων στη διαπραγμάτευση αυτού του ψηφίσματος. Αναλαμβάνουμε τις ευθύνε μας και επομένως είναι σειρά σας τώρα να σταθείτε κι εσείς στο ύψος ε, αυτής ε, της πρόκλησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σεζορνά. Ακολουθεί ο κύριος Μαριάννη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά την υγειονομική κρίση, η ε, έλλειψη προετοιμασία είναι θανατηφόρα και δεν θα πρέπει να καταγγέλουμε πλέον του εθνικισμού και του λαϊκισμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε στην αρχή ε, τη κρίση ότι δεν ήταν προετοιμασμένη. Δεν αρκεί το να ανύπτουμε τα σχήρι μα όταν τα συστήματα υγεία ε, ε, υποφέρουν και οι οικονομίε μα πάσχουν. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια εναλλακτική λύση. να πρέπει να αποφύγουμε όλες αυτές τις τις ιστορίες και υπάρχει και ο εφιάλτης ε, να στραφεί αλλού η προσοχή ε, του λαού διότι υπάρχουν πολλά άσχημα όνειρα εκεί. Επομένως ε, θα πρέπει να δούμε τα δόγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Γαλλία η κυβέρνηση παρουσιάζει ένα προϋπολογισμό ε, κοινωνικής ασφάλισης ο οποίος ε, πέφτει ακόμα και κάθε χρόνο και φέτος ε, θα έχουμε 4 δις ευρώ και ένα δις μόνο είναι για τις νοσοκομιακές υπηρεσίες. Τα 3 δις λοιπόν που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα κράτη-μέλη δεν αρκούν για να πληρώσουν τίποτα. Είναι ψυχία σε σχέση με τα, ο κόστος τα τελευταία χρόνια. Η Αυστρία και η Δανία προτείνουν δική του στρατηγική για να βγούμε από το lockdown και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει ένα ενοποιημένο σχέδιο, όχι για να καταπολεμήσουμε τον κορονοϊό, για να μην χάσει την αξιοπιστία τη. Η Γερμανία αποφασίζει να κλείσει τα σύνορά τη όταν ξεκινάει η κρίση, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπαρτύρεται για να υπερασπιστεί την ε, συνθήκη Σέγγεν. Όταν η ύφεση και η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση ε, θα χτυπήσει τι αγορέ εργασία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχρώνεται να αναστείλει όλου του κανονισμού για να μπορέσει να αναστείλει και την ύφεση. Τι θέλετε λοιπόν, έχετε ένα αρχιτεκτονικό οικοδόμημα το οποίο θα πρέπει ε, να το καταργούμε ε, σε κάθε κρίση. Θα πρέπει λοιπόν ε, να δούμε τι γίνεται, χωράμε στην προσχώρηση της Αλβανίας και της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πιέσεις για να αυξήσουμε τη συμβολή στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Οι λαοί θα δούνε όλους αυτούς που τους οδήγησαν σε αυτόν τον ε, ε, φιάλτη. Ε, πραγματικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα δούνε ότι υπάρχει προνομιακή πρόσβαση λόγω των ευρωπαϊκών κανόνων άλλων επιχειρήσεων στην περιοχή τους. Οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα θέματα ε, και να στηρίξουν ε, σε κοινωνικό επίπεδο και επομένω ε, θα δείτε ότι χρειαζόμαστε μόνο ε, αυτούς οι οποίοι σε εθνικό επίπεδο μπορούν να προχωρήσουν. Οι χώρες οι οποίες μπορούν να επιφορηθούν από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Αλληλεγγύης δεν μπορούν να το κάνουν διότι γνωρίζουν ότι δεν είναι οι λαοί που θα, το, θα αντιμετωπίσουν την αποτελεσματικότητα αλλά η διοίκηση των Βρυξελών. Θα πρέπει λοιπόν να συγκρατήσουμε τα μεταναστευτικά ρεύματα και ταυτόχρονα η ε, η υπηρεσία εξωτερικής δράσης φαίνεται ότι είναι μη αποτελεσματική στη Λιβύη και στην Τουρκία από όπου θα έρθουν την επομένη οι μετανάστες ε, του κορονοϊού. Πραγματικά λοιπόν η Ευρώπη ε, θα πρέπει να δει τι γίνεται. Δέχεστε να μας κατηδάσουμε στο θάνατο για να υποστηρίξουμε έναν ενιαίο νόμο. Για μένα λοιπόν δεν αναγνωρίζω ε, φίλο αυτός που απλώς του αρέσουν τα λόγια. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν να δει τι θα κάνει πραγματικά. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μαριάννη. Ακολουθεί για 1,5 λεπτό κύριο Τζαμπάτσκι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επίτροπε, συνάδελφοι, μέχρι στιγμής κανείς δεν είπε κουβέντα κατά της κομμουνιστικής Κίνας. Όλοι σιωπούν. Σιώψε και εκείνα, διέσπρεψέματα. Όπως πριν ε, λίγο καιρό, λίγα χρόνια είπαν ψέματα και οι Σοβιετικοί για το Τσερνομπίλ ε, με αποτέλεσμα χιλιάδες θύματα εδώ στην Ευρώπη. Κανείς δεν είπε τίποτα για τις ευθύνε που έχει η κομμουνιστική Κίνα. Δεύτερον, Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν αυτή που καθυστέρησε και λόγω αυτών των καθυστερήσεων τα κράτη-μέλη χρειάστηκε να κλείσουν τα σύνορά τους. Τρίτον, Αγαπητέ Σαλ Μισελ, προσφυλέστατε, θα έπρεπε να ντρέπεστε. Και πιστεύω ότι πρέπει να ντρέπεστε πραγματικά που σήμερα, εν μέσω όλων αυτών, αποφασίζετε σήμερα τη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες οδηγούς από την Ανατολική Ευρώπη, Βούλγαρους, Τσέχους και λοιπούς, οι οποίοι σώζουν ζωές ανθρώπινες ε, στη Δυτική Ευρώπη. Τώρα είναι ευπρόσδεκτοι, τώρα δεν σας πειράζει ο χρόνος ανάπαυσής τους ή αν κοιμούνται μέσα στα φορτηγά τους. Αύριο θα τους πετάξετε πάλι έξω με τις κλωτσιές. Τι υποκριτικό. Δεν είναι καν υποκρισία, είναι κάτι περισσότερο, είναι τρέλα. Για τους Ευρωπαίους συντηρητικούς, εμείς δεν πρόκειται να σας στηρίξουμε σε αυτή τη δήλωση. Σήμερα που χρειαζόμαστε λογικά οικονομικά μέτρα, αυτό το κείμενο έρχεται και μας πουλά ε, φανταστικά σενάρια και αν δεν δράσετε ε, υπεύθυνα θα ξανακατέληξουμε σε άλλο ένα Τσερνόμπιλ. Ε, ο κύριος ε, Μποτέγκα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Να ευχαριστώ τον κύριο Μισελ. Όπως συνήθως η... ακούμε ότι η λύση είναι περισσότερη αγορά. Όμως αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε ε, μια αγορά η οποία δεν μπορεί να παίξει το ρόλο της. Δεν είναι λέω μόνο ότι λείπουν μάσκες για αναπνευστήρες. Τα φάρμακα λείπουν. Λείπουν ε, ή τα εμβόλια. Πολλά από αυτά τα θύματα θα μπορούσαμε να τα είχαμε ε, αποφύγει εάν είχαμε τον εξοπλισμό. Δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζονται αυτά τα φαινόμενα. Γνωρίζαμε ότι χρειαζόμασταν μάσκες. Αλλά όλα βέβαια έχουν να κάνουν με το χρήμα. Οι πολυεθνικές προτιμούν να επενδύσουν αλλού. Είναι κοινικό αυτό. Όλοι θέλουν τώρα βέβαια θεραπεία, όλοι θέλουν εμβόλια και οι μεγάλες φαρμακευτικές είναι έτοιμες να πλώσουν τα χέρια τους και να μαζέψουν τα χρήματα με αποκλειστικά δικαιώματα, με πατέντες. Για μένα είναι σαφές αυτό. Δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα από αυτή την πανδημία. Θα πρέπει να αλλάξει να αλλάξει το σύστημα για να προστατέψουμε τις πατέντες θέλουμε υποχρεωτικές άδειε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να σταματήσουμε να έχουμε αυτές τις ιδιωτικές πατέντες, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Στην Νότια Αφρική οι πολυεθνικές δεν είχαν δεχτεί ε, να μειώσουν τα, το, τις τιμές των φαρμάκων για το AIDS και εκεί ο Νέλσον Μαντέλα το επέβαλε Θέλετε λοιπόν να είστε στο πλευρό της ζωής ε, ή ε, στο πλευρό των μεγάλων φαρμακευτικών εταιριών. Ευχαριστούμε τον κύριο Μποτέγκα. Ακολουθεί για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ κύριο Σκομίν Ολιβέηρες. Ε, όταν... Όταν εδώ στα Ιταλικά δεν ήξερα ότι πολύ σύντομα θα είχα και άλλο πολύ σημαντικό λόγο να ε, το κάνω εδώ. Είναι ένας ε, πάρα πολύ σημαντικός λόγος για να εκφράσω την αλληλεγγύη μου ε, στην χώρα που χτυπήθηκε περισσότερο από τον κορονοϊό, από αυτή την καταραμένη πανδημία. Διότι όπως όλες οι χώρες της Ιταλίας έτσι και η Καταλωνία πλήττεται από τον κορονοϊό. Σήμερα θα ήταν μια μέρα για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας σε κάθε γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι αυτή η οικονομική κρίση και οικονομική και κοινωνική ε, πλήττει όλε μα τι χώρε. Σήμερα περισσότερο από ποτέ η Ευρώπη θα πρέπει να θεωρήσει ότι είναι μια ενιαία κοινωνία και είναι η μέρα για να εκφράσουμε βεβαίω την αλληλεγγύη μα, τη δική μου την αλληλεγγύη και των ε, συντρόφου μα Ευρωβουλευτών, τον Κάρλο Πουτζεμόν και την Κλάρα Μπουλσεδίλ με το σύνολο τη ε, ισπανική ε, κοινωνία και φυσικά την αλληλεγγύη μα και τον πόνο μα για του θανάτου που προέκυψαν από αυτή την πανδημία. Ιδιαίτερα στην περιοχή τη Μαδρίτη και τη Λαριόχα. Θα πρέπει να έχουμε νέα και ισχυρά μέσα για να αντιμετωπίσουμε του βασικού στόχου αυτή τη κρίση, τη υγειονομική και τη οικονομική σε οικονομικό επίπεδο υποστηρίζουμε πλήρω την πρόταση να υπάρχει ένα ταμείο που θα χρηματοδοτηθεί από ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα υποστηρίζεται από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Σε υγειονομικό επίπεδο, φιλοδοξία για να δώσουμε αίθουσε σε στρατηγικέ ε, έρευνα και υγεία που θα μα επιτρέψουν να περιορίσουμε δραστικά το χρόνο που χρειάζεται για να βρεθεί αποτελεσματικό εμβόλιο για την πάταξη αυτή ή των μελλοντικών πανδημιών. Αν υπάρχει δημόσια πιο εύρωστη ε, έρευνα σε διεθνές και ε, παγκόσμιο επίπεδο θα μπορέσουμε να έχουμε αποτελέσματα. Ευχαριστούμε κύριε Κομίνη Ολιβέρες. Για δύο λεπτά ο συνάδελφος κύριος Μουρεσάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η εμπειρία των τελευταίων δύο μηνών, ε, συναδελφοί, δείχνει ότι κανένα κράτο μόνο του δεν μπορεί να νικήσει αυτό τον ιό. Η δική μα απάντηση, η ευρωπαϊκή απάντηση, ήδη έκανε μεγάλη διαφορά σε πολλά μέρη ε, δείξαμε ότι η αλληλεγγύη νικά του εγωισμού και ότι μπορούμε να βοηθήσουμε του ευρωπαϊκού λαού. Πριν τρει εβδομάδε ε, σταθήκαμε εδώ και αποδεσμεύσαμε 37 δισεκατομμύρια ευρώ για την καταπολέμηση του κορώνα. Και εδώ σε αυτή την αίθουσα ρώτησα εγώ τον ε, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορείτε να κάνετε περισσότερα, χρειάζονται περισσότερα και τη ζήτησα να δώσει ε, οτιδήποτε υπάρχει από αποθεματικά που αχρησιμοποιητά για τον προπολογισμό του 2020 για να χρησιμοποιηθούν για την καταπολέμηση του κορονοϊού. Και αυτό προτείνει τώρα η Κομισιόν. Πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ να αποδεσμευτούν για του ανθρώπου που τα έχουν ανάγκη. Πρέπει να το εγκρίνουμε και γρήγορα για να γίνει νόμο και να φτάσουν τα χρήματα αυτά σε όσου θα χρειάζονται, στου ασθενεί, στου γιατρού, στα νοσοκομεία. Αλλά εγώ λέω χρειάζονται περισσότερα ακόμα. Αυτή δεν είναι παρά η αρχή. Πρέπει να προγραμματίσουμε και για το μέλλον, συνάδελφοι. Η Ευρώπη πρέπει να βοηθάει εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, στα νοσοκομεία. Βλέπουμε χώρε, περιφέρειε, πόλει που δεν καταφέρνουν να σώσουν τις ζωές των πολιτών τους. Οι άνθρωποι έχουν στραμμένο το βλέμμα προς εμάς για λύσεις. Και εγώ λέω, έχω ένα σχέδιο, έχω μια πρόταση. Ας δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό υγειονομικό ταμείο που θα βοηθήσει τα νοσοκομεία σε κάθε γωνιά της Ευρώπης. Εγώ προτείνω να δημιουργήσουμε ένα ταμείο 50 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα βοηθήσει να βελτιωθεί η κατάσταση σε όλα τα νοσοκομεία, σε όλη την Ευρώπη για να μπορέσουμε να είμαστε βέβαιοι ότι όλοι οι άνθρωποι όποιοι και να ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνουν σωστή υγειονομική περίθαλψη. Το ερώτημα είναι υπάρχουν τα χρήματα και η απάντησή μου είναι φυσικά και τα έχουμε. Θα πρέπει να στείλουμε τα χρήματα αυτά όπου υπάρχει μεγάλη ανάγκη για να σώσουμε τις ζωές των πολιτών της Ευρώπης. Η ομάδα μου το προτείνει αυτό ως τροπολογία σήμερα για το ψήφισμα και εγώ ζητάω από όλες τις ομάδες να συνενωθούν πίσω από αυτό το στόχο. Το έργο αυτό θα πρέπει να γίνει έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του 2020 θα πρέπει να το θυμόμαστε γιατί δημιούργησε ένα ευρωπαϊκό υγειονομικό ταμείο που έδωσε ελπίδα στους λαούς της Ευρώπης και έσωσε ζωές. Ευχαριστούμε κύριε συνάδελφε Μουρεσάν για 2,5 λεπτά για 1,5 λεπτό συγγνώμη συνάδελφος Μουρενό Σάντσες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Απέναντι στην κρίση η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να δώσει μια απάντηση η οποία να μην είναι τολμηρή. Φτάνει πια με τα οικονομικά δόγματα. Απέναντι αυτή την ιστορική πρόκληση, η Ευρώπη πρέπει να δείξει πολιτικό θάρρο, αλληλεγγύη, καινοτομία για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτήν την κοινωνική και οικονομική κατάσταση, χωρί να μείνει κανεί πίσω εδώ κινδυνεύει το κοινό μα μέλλον. Η συμφωνία του Eurogroup είναι ένα πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά δεν αρκεί. Η Ευρώπη χρειάζεται ένα συνολικό σχέδιο ανοικοδόμησης, φιλόδοξο, μεσομακροπρόθεσμο, ένα νέο σχέδιο Marshall ευρωπαϊκών επενδύσεων, κοινό, Όπω πρότεινε ο πρόεδρο Σάντσεθ. Ένα σχέδιο που να προβλέπει κάποια μέσα όπω ε, τα ευρωομόλογα που να διέπονται από αλληλεγγύη. Πρέπει να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα προ όλου του πολίτε σήμερα, να εγκρίνουμε ένα πρώτο δικό χάρτη, το αυτό το κοινό ψήφισμα που θα, υποστηρίξουν, που θα υποστηρίξει την μου και μια σειρά από δημοσιονομικά και ρυθμιστικά μέτρα που θα έρθουν να απαντήσουν στι υγειονομικέ, οικονομικέ και κοινωνικέ ανάγκε των συμπολιτών μα, ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων θα πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου το κοινό συμφέρον, το κοινό όφελο. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα οικονομικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μα και ό,τι προβλέπεται στη συνθήκη. Θα το κάνουμε αυτό υπερασπιζόμενοι τη δημοκρατία, το κράτο δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Θα πρέπει η ανάκαμψη να έχει στο κέντρο τη την ψηφιακή μετατροπή, ε, το Green Deal, τον διατροφικό τομέα, τον τομέα τη ε, ε, γεωργίας της αλίας. Θα πρέπει λοιπόν να συμμετάσχει και αυτό το Ευρωκοινοβούλιο στην προπαρασκευή αυτού του σχέδιου ανάκαμψης να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας. Ευχαριστούμε κύριε Μωρινό Σάντσες. Κύριε συνάδελφε Σάντσες, ε, είχατε 1,5 λεπτό. Έχει περάσει το 1,5 λεπτό σας. 1,5 λεπτό είχατε. Συγγνώμη, δεν σα έδωσα ξανά το λόγο. Είχατε το λόγο για 1,5 λεπτό και έχετε περάσει τα δύο ήδη. Είναι θέμα σεβασμού προς τους συναδέλφους σας και σεβασμού προς όσους μας ακούνε έξω από αυτό το κοινοβούλιο να ακούσουν όλοι έγκαιρα και να μπορέσουν να ακούσουμε και τα σχόλια του Επιτρόπου στο τέλος της συζήτησης για να προλάβουμε. Ακολουθεί η συναδέλφος κυρία Ρης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο COVID-19 έρχεται να δείξει το καλύτερο αλλά και το χειρότερο της ανθρώπινης φύσης και το καλύτερο είναι αυτή η συμμετοχή, η αυταπάτνηση χωρίς όρια ε, των, ε, του ιατρικού προσωπικού και όλες αυτά, όλα αυτά τα ε, οι κινήσεις αλληλεγγύης παντού στον κόσμο ε, κάποιοι που ξαφνικά μαθαίνουν να ράβουν για να μπορέσουν να φτιάξουν μάσκες προστασίας, οι ίδιοι αυτοί οι πολίτες οι οποίοι με τον παραδειγματικό τους, ε, πραγματική τους δράση μας εμπνέουν και εμά και μας λένε τι κάνει τελικά η Ευρώπη, κάνει αρκετά, γιατί οικονομικά ελέγχθησαν ήδη πολλά. Το μέλλον θα μας δείξει τι θα γίνει με το σύμφωνο σταθερότητας, κρατικές ενισχύσεις, ε, ε τα ταμπού πραγματικά αυτή τη στιγμή τα ξεπερνάμε. Το Κοινοβούλιο ζητάει περισσότερα σήμερα. Ε, ζητάει ε, πλέον αυτά τα κορονομόλογα, τα λέγγια ομόλογα, ε, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την καταστροφή που δημιουργεί αυτή η κρίση. Η οικονομικό επίπεδο βεβαίω είναι πολλά τα ερωτηματικά και δεν πρόκειται επάπειρον να κρυβόμαστε πίσω από τα όρια τη συνθήκη. Δεν το καταλαβαίνει κανείς αυτό. Τι έκανε τελικά το CDC σε επίπεδο πρόληψη, σε επίπεδο προετοιμασία, γιατί με το εύρο τη κρίση αυτή, η Κομισιόν δεν ξεκίνησε την ανθρωπιστική βοήθεια στο, στο ιστορικό της για να βοηθηθούν τα νοσοκομεία στη Μιλούζ, στον Πέργαμο, ε, στην ε, Μαδρίτη. Τι έγινε με το Ευρωπαϊκό Ιατρικό Σώμα. Έχουμε τα μέσα. Αυτό που μα έλειψε είναι το θάρρο. και θέλω να πω κάτι και αφήστε με να τελειώσω γιατί είναι πολύ σημαντικό ήθελα να μιλήσω για τους ηλικιωμένου, οι οποίοι πληρώνουν το πιο μεγάλο τίμημα ένα στους τρεις νεκρούς στη Γαλλία ένα στους δύο στο Βέλγιο ήθελα να πω στην κυρία Φοντελάιν που δεν είναι πια εδώ όμως ότι το να καταδικάζουμε τους ηλικιωμένου σε πολλούς μήνες εγκλισμού δεν είναι η σωστή λύση. Να γίνουν τεστ, να, υπάρξουν, να δοθούν μάσκες. Δεν έχω τη λύση να τη δώσω εγώ σήμερα, αλλά δεν μπορούν οι ηλικιωμένοι μας ε, να ζουν σε αυτήν την ε, απομόνωση, σε αυτήν την ε, δυστυχία. Πρέπει να τους στρέψουμε ένα χέρι βοδού. Ευχαριστούμε κύριε Ρης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο, κύριος Ντεμάν για ένα λεπτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Τον Ιανουάριο όταν ε, μάθαμε ότι υπήρχε ε, ένας ε, θανατηφόρος ε, ιός στην Κίνα δεν ε, έλαβε κανένα μέτρο για τους ανθρώπους που έρχονταν από την Κίνα. Δεν υπήρχαν τον υπαρχή αριθμό ελέγχων, ήταν ανοιχτά τα σύνορα, ορθά ανοιχτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τις 20 Μαρτίου, δεν εξέτασαν πώς θα μπορέσουν να προστατεύσουν τους διάφορους κλάδους, δεν ασκήθηκε επαρκής πίεση για να κλείσουν οι αγορές αυτές οι ζωικές ε, στην Κίνα και δεν εξέτασαν προσεκτικά τι γίνεται στα εργαστήρια της Βουχάν,